Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12.30. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε την έκθεση του François Αλφονσί για την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο. Να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, ο οποίος έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η έκθεση για την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και τις τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον κυρίως στην Μεσόγειο εδράζεται σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, τον προγραμματισμό 2014-2020 ως προς την ε, πολιτική του Ταμείου Συνεχής και την πολιτική για τις περιφέρειες και ως προς την ε, ε, ε, ως προς την, ε, στις μακροπεριφέρειες οι οποίες έχουν ε, ήδη συσταθεί. Το άλλο στο οποίο σε βασίζεται η έκθεση αυτή είναι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η κρίση χρέους, οι πολιτικές εξελίξεις στις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αραβικές χώρες από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Ζητώ συγγνώμη μισό λεπτό να βρω το έγγραφο της ομιλίας μου, ζητάει ε, ομιλητής. Elle Και έτσι πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό αναφέρεται στα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την πολιτική γειτονία, ε, το προτεξιακό καθεστώς και έτσι μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία μεγαλύτερου συντονισμού και διαβούλευσης για τα έργα που θα γίνουν στο μέλη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα ε, γνωρίζουμε για το μέλλον. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη στρατηγική του Ιωνίου, η οποία καλύπτει την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Όλα αυτά είναι κάποια πρώτα βήματα πολύ σημαντικά. Και στη Δυτική Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται τέτοια διαβήματα και καλύτερο συντονισμό θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση του συνόλου του μεσογειακού χώρου. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και τα θέματα εδαφικής συνεργασίας, η εδαφική συνεργασία γενικότερα είναι ένα εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες στηρίζεται στον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Δεν μας χρειάζονται περισσότερες ή νέες πιστώσεις, μας χρειάζονται νέα και πιο καινοτόμα έργα και θα πρέπει να εμπλέκονται οι τοπικοί παράγοντες, η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να έχουμε σωστή διαχείριση σε πολλαπλά επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει την πραγματογνωμοσύνη της, την εμπειρία της και ε, στο θέμα αυτό και θα πρέπει να το προωθήσει και η Κυπριακή Προεδρία τους επόμενους ε, μήνες. Έχουμε βούληση να συνεργαστούμε γύρω από αυτό το εγχείρημα μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε όλο το μεσογειακό χώρο. Πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, να στείλουμε ένα θετικό πολιτικό μήνυμα για το μέλλον, για ένα μεσογειακό χώρο ο οποίος πλήττεται από την οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή στο σύνολό του. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους συναδέλφους μου από την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όλους όσοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους ε, για την την έκθεση αυτή. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή για τον Πολιτισμό και από την Επιτροπή για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, τον κύριο Σαλαβράκο πιο συγκεκριμένα για τη δουλειά που έκανα και για το ότι εμπλούτησε την έκθεση που σας παρουσιάζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε πέντε ομιλητές που ζήτησαν το λόγο και πέντε λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Να ξεκινήσουμε με κάποιον ο οποίος ε, παίρνει για πρώτη φορά το λόγο, την κυρία Μπεναράπ Αρτουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι μέσα στο ένα λεπτό που έχω στη διάθεσή μου σε αυτό που είπε ο κύριος Αλφόνση. Είμαι συγγήτρια για γνωμοδότηση εξ μέρου Επιτροπή ε, Παιδεία. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική ανοίγει ιδιαίτερε προοπτικέ ε, στον ε, τομέα τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Μου φαίνεται ότι πρόκειται για ένα σωστό πλαίσιο για την προβληματική αυτή τη περιοχή που τα γεγονότα των τελευταίων ετών θα πρέπει να μα ενθαρρύνουν να απτύξουμε μια πολιτική γειτονία. Θα ήθελα να επιμείνω προς τρία σημεία. Καταρχάς, η συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιουργώντας συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Νεολαίας, που θα πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστό. Δεύτερο, Δημιουργία δικτύων μεταξύ των ευρωπαϊκών παρεπιστημίων και άρση των εμποδίων για την κυκλοφορία των ερευνητών, των φοιτητών και των, των σπουδαστών και των ε, καθηγητών με ε, παροχή θεωρήσεων. Τρίτον, η ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας σε αυτό το δίκτυο μέσω της χρηματοδότησης και της στήριξης των προγραμμάτων του προγράμματος Εράσμους και παρέχοντας αυτομάτως θεωρήσεις σε τους ανθρώπους αυτούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλφοσί για την συνεργασία του καθώς και στους συναδέλφους που συνετέλεσαν στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Καρό. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της μακροπεριφερειακής στρατηγικής και το γεγονός ότι θα πρέπει να βασίζεται στη διακυβέρνηση όπου θα εμπλέκονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αλλά θα υπάρχει και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των πανεπιστημίων και στη διαδικασία εφαρμογής και στη διαδικασία σχεδιασμού αυτών των στρατηγικών για να υπάρξει μια τέτοια σωστή εφαρμογή θα πρέπει να εστιαστούν τα ε, ε, προγράμματα των χωρών μελών στις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής. Ζητάμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν ε, τους στόχους της περιοδικής διαδικασίας ελέγχου. Το 2010 το Κοινοβούλιο ζήτησε να δοθούν 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τις προπασκευαστικές δράσεις που είχαν στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Αλφονσί για την ε, έκθεση που μας παρουσιάζει, αλλά και όλη την ε, προεργασία που έγινε, τη διαβούλευση με εθνικές και τοπικές αρχές από ολόκληρη την μεσογειακή λεκάνη από το βορρά και το νότο. είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το ότι συζητούμε για μια συγκροτημένη ε, ε, στρατηγική μακροπεριφερειών διότι χωρίς πρόσθετους πόρους δίνεται μια προστιθεμένη αξία στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές πολιτικές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Ε, έχει μπει σε ένα δρόμο πια και πιστεύω ότι γρήγορα η Επιτροπή θα απαντήσει θετικά μαζί με μια συγκεκριμένη στρατηγική ε, που θα δώσει ε, δυνατότητα ανάπτυξης των πρωτοβουλειών. Είναι ε, σημαντικό ότι στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και μια ναυτιλιακή διάσταση και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και εκτός της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Τέταρτος, ο, τέταρτη ομιλήτρια, η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες είναι πολύ ευεργετική, διότι δίνει νέες προοπτικές στα διάφορα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει το καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και έτσι επιτυχάνονται πιο εύκολα οι στόχοι για την Ευρώπη του 2020. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η στρατηγική για τη θάλασσα της Βαλτικής και την μακροπεριφέρεια αυτή. Ε, υπάρχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες και στη Νότια Ευρώπη επίσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας στην ε, περιοχή. Η χάραξη στρατηγικής μακροπεριφερειών, μακροπεριφέρειας στην Μεσόγειο είναι ένα βήμα προς τα μπροστά μεταξύ χωρών που μοιράζονται, που έχουν παρεμφερεί ιστορία, κοινό πολιτισμό και κουλτούρα και έτσι μπορούν να βελτιώσουν ε, τις συνθήκες ζωής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον ε, Επίτροπο κύριο Κάλλας, μιλήσατε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εταιρική σχέση προς την Ανατολή. Ελπίζω να επιδείξετε το ίδιο ενδιαφέρον και στη συζήτηση για τον Νότο. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιότιμα Μέλη ευχαριστεί τον κύριο Αλφονσί για την ε, ε, έκθεση του αυτή και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πόσο ε, μεγάλο είναι το πολιτικό ενδιαφέρον για μια στρατηγική στη Μεσόγειο και λαμβάνει υπόψη της βεβαίως και τις πολύ σημαντικές πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν και πολιτικές δυσκολίες. Η στρατηγική που προτείνει ο κύριος Αλφονσί, δηλαδή δυτική, κεντρική και ανατολική, περιλαμβανομένη στι θάλασσε της Αδριατική και του Ιωνίου Πελάγους, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική που θα πρέπει να αντιληφθεί περαιτέρω. Αυτοί οι τρει άξονε δηλαδή. Ειδικότερα όσον αφορά στην πρωτοβουλία Αδριατική και Ιωνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πάντες να αντλήσουν τα διδάγματα Τη στρατηγικής μακροπεριφέρειας που έχουμε ήδη για τη θάλασσα της Βαλτικής και για τον Δούναβη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει όποια πρωτοβουλία προκύπτει η οποία κάνει τις χώρες και τις περιφέρειες να συνεργαστούν ακόμα περαιτέρω είτε με την τρέχουσα μορφή είτε με τη μορφή της μακροπεριφέρειας. Αυτή είναι και η πιο καλή λύση. έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2011, όπου καλούνται τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση όλων αυτών των στρατηγικών μακροπεριφερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει κάθε πρόοδο που μπορεί να σημειωθεί ε, στο πλαίσιο της περαιτέρω μεσογειακής συνεργασίας. Τώρα, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος σίγουρα χρειάζεται εντολή που να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο για να δημιουργηθεί αυτή η μακροπεριφέρεια και η στρατηγική για την εκάστοτε μακροπεριφέρεια. Και όλοι βέβαια γνωρίζετε ότι πολύ συχνά, ειδικότερα σήμερα, εξετάζονται ε,